τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΥΠΑ της εκπροσώπου ε, όσον αφορά ε, τη ρήτρα για την αμοιβαία συνδρομή άρθρο 4270 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η κυρία Μογκερίνη έχει ξανά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν είναι απλή η κατάσταση για την Ευρώπη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε άνευ προηγουμένου προκλήσεις. Οι συμπολίτες μας ε, μας ρωτούν ποιο είναι το νόημα της Ένωσης η Ένωση των 28 είναι εξαιρετικά περίπλοκη και πλουραλιστική, υπερβολικά πλουραλιστική για να μπορέσει να λάβει αποφάσεις σε αυτές τις τόσο δύσκολες καταστάσεις. Απάντησή μας ε, απέναντι στις επιθέσεις του Παρισιού εξέπληξε πολλούς παρατηρητές. Είχαν σκεφτεί πολύ ότι σε αυτές τις σκοτεινές ώρες η Ευρώπη θα διαλυόταν, θα ξεσκιζόταν από εσωτερικές διαμάχες. αυτό το θέμα το μας απασχόλησαν σε όλα τα συμβούλια μετά από τις 13 Νοεμβρίου. Η απάντησή μας ήταν αυτή μιας πραγματικής ένωσης όμως. Όπως γνωρίζετε, μετά τις ε, τρομοκρατικές ρυθμίσεις η Γαλλία ζήτησε την αρρωγή της των άλλων κρατών μελών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 17 Νοεμβρίου, μετά από το Συμβούλιο ε, Κορυφής, τα κράτη-μέλη έστειλαν έντονο μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς τη Γαλλία. Πέρα από το πολιτικό μήνυμα, το άρθρο 42.7 της Συνθήκης συμπεριλαμβάνει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη. Και όντως τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση θα παρέχουν βοήθεια και αρρωγή στο κράτος μέλος που δέχεται επίθεση με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτή η διατύπωση συνήθως γίνεται νοητή ως χρήση στρατιωτικών μέσων, αλλά αναμφίβολα το 42.7 καλύπτει επίσης την αρρωγή μέσω άλλων ε, εργαλείων ή μέσων στήριξης μη στρατιωτικής φύσης. Το άρθρο αυτό εκφράζει ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης και εξαρτάται από το κράτος μέλος να ορίσει την ακριβή φύση της βοήθειας ή της αρρωγής που τελικά θα προσφέρει. Το πλαίσιο είναι ευρωπαϊκό. Η βασική αρχή είναι ενότητα μέσα στην αντικσότητα. Η Γαλλία ζητά στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά ενωμένη. Ο Γάλλος Υπουργό Άμυνας υπέβαλε δύο συγκεκριμένα αιτήματα προς τους υπουργούς. Πρώτον, να στηρίξουν επιχειρήσεις που θα κάνει η Γαλλία κατά τον ΤΑΕΣ στη Συρία και στο Ιράκ και δεύτερον σε να καλύψουν ε, την έλλειψη πόρων που μπορεί να προκύψουν σε στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της γαλλικής επίθεσης κατά του ΤΑΣ. Η Γαλλία προσέγγισε το κάθε κράτος μέλος διημερός με συγκεκριμένα αιτήματα μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αμήνης αλλά επίσης ε, και μέσω των δομών για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες όπως γνωρίζετε για την εφαρμογή του άρθρου 42.7 και όπως γνωρίζετε το άρθρο αυτό ποτέ δεν το είχε κανείς επικαλεστεί μέχρι στιγμής. Η εφαρμογή του λοιπόν μπορεί να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Και ενώ το άρθρο 42.7 δίζει συγκεκριμένα το ρόλο των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέσα και οι μηχανισμοί του μπορεί να υπάρξουν για να αντιμετωπιστούν οι απειλές προς τα κράτη-μέλη. Ακόμα και αν λοιπόν δεν ορίζεται συγκεκριμένα στη διατύπωση του άρθρου αυτού της συνθήκης, εμείς στο Συμβούλιο μετά το αίτημα της Γαλλίας συμφωνήσαμε στο να ε, αναμειχθούν ή να εμπλακούν οι ευρωπαϊκές δομές στην ε, ε, ανάλυση αυτών των διατάξεων και βέβαια ε, να συντονίσουμε οποιοδήποτε αίτημα που μπορεί να έχει αντίκτυπο στις ε, επιχειρήσεις ε, της ευρωπαϊκού επίπεδου. Έτσι και η Γαλλία έδωσε, προσέφερε ενημέρωση τόσο στην Στατιστική Επιτροπή όσο και στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου. Οι γαλλικές ενέργειες κατά του ΝΤΑΕΣ μέχρι στιγμής δεν είχαν επιπτώσεις στις ε, ευρωπαϊκές αποστολές και επιχειρήσεις εκεί που η Γαλλία δηλαδή δραστηριοποιείται. Βεβαίω η Γαλλία μπορεί ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσέξει και σε άλλες συμπληρωματικέ συνεργασίες ε, αν αυτό χρειαστεί. Οι δεσμεύσει και οι συνεργασίες θα είναι σύμμορφες με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το, σύμβαση του ΝΑΤΟ για τα κράτη-μέλη που είναι μέλη του. Σήμερα όλοι συνειδητοποιούμε πως δεν υπάρχει κράτος, έθνος μόνο το που μπορεί να ε, σταθεί απέναντι σε αυτές τις απειλές. Αυτή η ενότητα που αισθανόμαστε είναι αυτή που είναι και η δύναμή μας. Η ο συγκεκριμένος χαρακτήρας των εξωτερικών μας πολιτικών δεν είναι παθητικό μας. Αποτελεί την ισχύ της Ένωσης. Καμιά άλλη δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να κινητοποιήσει τόσο μεγάλη ποικιλία ε, μέσων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Η Ένωση μέσα στη διαφορά. Αυτή είναι η δύναμή μας, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε χωρίς να φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις διατάξεις της συνθήκης όταν και εφόσον εξυπηρετούν εθνικά ή ε, συλλογικά συμφέροντα. Συχνά διαμαρτυρόμαστε για τις ε, διχόνοιές μας, για τις διαφορές μας, όμως ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει αυτή τη φορά περίφωνος η ενότητα σε αυτήν την συγκεκριμένη περίσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε Μογκερίνη. Ξεκινάμε με τη συζήτηση για δύο λεπτά. Πρώτος ο κύριος συνάδελφος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Γαλλία ως πρώτη χώρα μετά από τα, τις φρικαλές επιθέσεις στο Παρίσι ζήτησε να λειτουργήσει η ρήτρα συνδρομής. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο και ως ομάδα του ΕΡΚ χαιρετίζουμε την σαφή υποστήριξη, ανεπιφύλακτη υποστήριξη της Γαλλίας. Γνωρίζουμε όμως από την άλλη πλευρά επίσης ότι αυτό το άρθρο συνδρομής κατά πρώτο λόγο είναι πολιτικό ζήτημα και ότι η κατάσταση για τη χώρα που πρώτη, ως πρώτη δημιούργησε αυτό το προηγούμενο δεν είναι καθόλου άνετη και ευχάριστη. Η ίδια η Γαλλία πρέπει ίδια να μεριμνήσει να καθορίσει τι χρειάζεται ακριβώς και να προσεγγίσει τα άλλα κράτη ώστε να βοηθηθεί. Εμείς ως Κοινοβούλιο στην δική σας προδιάδοχο το 2012 νομίζω ήταν ζητήσαμε πρακτικά μέτρα και κατευθυντήριες γραμμές να προτείνει σε περίπτωση που χρειαζόταν να λειτουργήσει αυτό το άρθρο συνδρομής και να εξετάσουμε πώς θα αντιδρούσαμε άμεσα. Ποιος, γιατί πράγμα θα ήταν αρμόδιος. Δυστυχώς μέχρι σήμερα όμως δεν συνέβη αυτό, δεν έγινε αυτό, το είπατε και εσείς οι ίδια εξάλλου. Και έχουμε και πάλι μια κατάσταση που βιώσαμε όπου τα σύνορα μεταξύ εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής ασφάλειας διαλύονται, είναι ασαφή και γι' αυτό για τις δυνατότητες ε, της συνθήκης όπως προσφέρονται για να δρομολογηθεί το άρθρο συνδρομής ε, για την εσωτερική ασφάλεια είναι προφανές ότι οι αστυνομικές αρχές, ε, οι τελωνιακές αρχές, οι σε πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους πρέπει να τις γνωστοποιούν, να υπάρχει αμοιβαία ενημέρωση, να μην περιμένουμε να συμβεί κάτι για την εξωτερική ασφάλεια. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται στενά μεταξύ τους και να το κάνουν αυτό και όσοι θέλουν να εμπλακούν σε αυτό πρέπει να μεριμνήσουν και να το πράξουν αυτό μέσω της δραστηριοποίησης της διαθρωμένης συνεργασίας, μόνιμης διαρκούς διαθρωμένης συνεργασίας ώστε να μπορέσει να αναλυφθεί κοινή δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Γκάλερ. Στην αρχή ξέχασα να αναφέρω, μια και υπήρξε αλλαγή, ότι έχουμε τέτοια πίεση που δεν θα έχουμε μπλε κάρτες στη συζήτηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω του ότι πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος. Για δυόμιση λεπτά τώρα ο συνάδελφος κύριος Πάσκου. I can only regret. Μπορώ να εκφράσω μόνο τη λύπη μου, διότι η έκθεση που ετοίμασα το 2012 ετοιμάστηκε τέσσερα χρόνια νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Έχοντας ακούσει αυτά που είπατε, δεν θα επαναλάβω αυτά που ζητούσαμε στην έκθεση. Ε, που έμειναν αναπάντητα αυτά που θέσαμε. Ο κ. Βαν Όρντεν, ο Τζόφρι γνωρίζει την ιστορία της ε, έκθεσης. Ε, δυστυχώς η έκκληση αυτή αγνοήθηκε. Συνεπώς όταν η Γαλλία επικαλέστηκε το άρθρο 222 που ρητά ασχολείται με την τρομοκρατία, το άρθρο 42.7, πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε δημιουργώντας προηγούμενο για μελλοντικές παρομοιες καταστάσεις σαν ε, πρώην Υπουργό Αμήνη, ε, βλέπω ότι υπάρχει πλεονέκτημα να προχωρούμε σαν αρχαρτογράφητα ύδατα, αλλά το σημερινό προηγούμενο που δημιουργούμε θα αρκεί αύριο σαν λύση. Η κατάσταση δείχνει για μια ακόμη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά διολυσταίνει προ δικό τη κόσμο. Όλο και περισσότερο διαχωρίζεται από την πραγματικότητα Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, πήραμε το Θεωρήσαμε ότι δεν θα επικαλεστούμε 42-7 ποτέ και δεν χρησιμοποίησαμε τα διπλωματικά σα αμυντικά εργαλεία όποτε χρειαζόταν και πρέπει να προσφύγουμε στη διαχείριση κρίσεων και περίπλοκε ε, λύσει που είναι και πιο δαπανηρέ για να αντιμετωπίσουμε τη σύγκρουση που έχουμε στο, στη θύρα μα στον κόσμο επικρατούν οι ε, πολιτικές ισχύω. Και δεν μπορούμε εμείς να μην χρησιμοποιούμε στατιστική ισχύ για να αμυνθούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται επίθεση χωρίς να έχει λύσει τα εσωτερικά της προβλήματα και η ανταπόκρισή της δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε ήπια δύναμη. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να αγνοεί τις πραγματικότητες, την πραγματικότητα που την περιλαμβάνει, περιβάλλει θα υποφέρει την ίδια μοίρα όπως και η κοινωνία των εθνών τη δεκαετία των 30. Κάτι που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Πάσκου. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος κύριος Φανόρδεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εστιαζόμαστε στην καταπολέμηση τη πραγματικά τρομοκρατική απειλή και να βοηθήσουμε τη Γαλλία και άλλου στενού συμμάχου οι οποίοι δέχτηκαν τρομοκρατικέ επιθέσει προσφάτω και να μην θέλουμε να προωθήσουμε αμυντικέ φιλοδοξίε που δεν έχουν θέση τη Ευρωπαϊκή Ενώση και θέλουν οι φεντεραλιστέ να τι προωθήσουν. Η ομάδα του ECR είναι κάθετα αντίθετο όσον αφορά το ψήφισμα που δειχνά διαθρωμένη ε, άμυνα, τη δημιουργία μονίμου αρχηγείου ε, τη Ευρωπαϊκή Ενώση συλλογική άμυνα άμυνα και να κινηθούμε προ αυτόνομη ένωση αμυντική εξορισμού που ήταν διαχωρισμένη από το ΝΑΤΟ. Είναι επικίνδυνε ανοησίε αυτά. Το καταλαβαίνουν οι ρεαλιστέ, πάρα πολύ καλά αυτό. Ε, προειδοποιούσαμε επί καιρό για του κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειγνύεται στην άμυνα. Αυτό μόνο πρέπει να είναι ει βάρο τη εθνική κυριαρχία και του ΝΑΤΟ η απαραίτητη αυτή συμμαχία που είναι αξιόπιστη για τους εχθρούς μας και η οποία καθησυχάζει τους συμμάχους. Πολλοί απογοητεύτηκαν ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα συμπεριλαμβάνεται η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή, διακοσμητική μίμηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, χωρί καμία βάση όμω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δυνατότητα να παράσχει συλλογική άμυνα. Εν πάση περιπτώσει, 22 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και το υπόλοιπο, το μικρό, με μία εξαίρεση, έχουν συμμετάσχει κατά κάποιο τρόπο σε δραστηριότητε του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να συμπεριληφθεί το άρθρο 7. Ε, συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, και σίγουρα δεν θα πρέπει να επικληθεί. εκτό βεβαίω, ο στόχο σα είναι να είσαστε προκλητικοί ή θέλετε σκόπιμα να δείτε το ΝΑΤΟ να βγει στο περιθώριο. Ευχαριστούμε συνάδελφε Βανόλεν. Για δύο λεπτά στη συνέχεια συνάδελφο Σπάιτα. Ευχαριστώ πολύ για την χρήση της ρήτρας συνδρομής από τη Γαλλία μας έδωσε μια ευκαιρία αλλά και υποχρέωση να καθορίσουμε το πλαίσιο και τους στόχους της. Η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή μα δίνει μια μοναδική ευκαιρία να λιάνουμε το έδαφο για μια ισχυρή αμυντική ένωση και έτοιμη να αντιμετωπίσει τι προκλήσει μέχρι σήμερα ερμηνευόταν ως διμερής υποχρέωση μεταξύ κρατών να βοηθούν εκείνο το κράτος το οποίο χρήζει βοηθείας. Πρέπει να βεβαιωθούμε όμως ότι θα υπάρχει ένα ορθό, σωστό πρόγραμμα δράσης, ώστε όλοι να κατανοούν τις υποχρεώσεις τους όταν ένα κράτος αποφασίζει να κάνει χρήση αυτού του άρθρου. Ένα κράτος που έχει ανάγκη πρέπει άμεσα να μπορεί να τύχει αυτή τη βοήθεια από τους υπόλοιπους. Ο χρόνος έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό δεν υποκαθιστά το άρθρο 5 της αμοιβαίας συνδρομής του ΝΑΤΟ που αφορά την απειλή εναντίον ενός κράτους οπότε πρέπει τα άλλα να συνδράμουν <clears throat> αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες απειλές από την τρομοκρατία και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε πολλές πτυχές που είτε είχαν αμεληθεί είτε δεν ε, ελήφθησαν υπόψη. Και τώρα, σε σχέση με το Σέγγεν, τα κράτη κλείνουν τα σύνορά τους και είναι έτοιμα να κατεδαφίσουν την ελευθερία κυκλοφορίας επί της οποίας θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενδυναμωθεί. Να μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες με ευφυή τρόπο για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Για να μπορέσουν τα δίκτυα πληροφοριών να λειτουργήσουν, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών ή τουλάχιστον να μπορεί η Ευρωπόλ να μπορει η να εχει περισσότερες αρμοδιότητες ώστε de facto να μπορεί να υλοποιεί ε, το εγκάσια και ε, διαδικτυούμενα ε, πλαίσια δράσης μέσα από αυτή τη δικτύωση και να υπάρξουν αυτές οι, αυτά τα πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Πάτς. Τώρα για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Κόλσο Περμούη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, απορρίπτουμε την δρομολόγηση αυτής της αμοιβαία ρήτρα συνδρομής, διότι η απάντηση θα ήταν δυσανάλογη. Θα ε, ρίχναμε λάδι στη φωτιά και έτσι θα υπήρχε πρόβλημα. Διαφωνούμε απόλυτα με την ερμηνεία που δίνει η Γαλλία. Όσο και υπάρχει η προσπάθεια αυτή, μια τρομοκρατική επίθεση δεν είναι πολεμική πράξη. Μια τέτοια ερμηνεία υπονομεύει το διεθνές δίκαιο, εξαπατώντας τις αρχές. Εδώ έχουμε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Πολιτικές δράσεις πρέπει να αναλαμβάνονται. Αστυνομικές δράσεις, δράσεις υπηρεσιών πληροφοριών, διακοπή χρηματοδότησης και μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου δεν μπορούμε να απεμβολήσουμε και να χάσουμε τις ελευθερίες μας. Δεν μπορούμε να σκοτώνουμε μύγες με κανόνια. Εδώ είδαμε ότι οι καταστράφηκαν κοσμικά κράτη με ε, εκατομμύρια ε, νεκρών και εκατοντάδες ε, χιλιάδων προσφύγων δημιουργώντας ένα τέρας όπως το Ντάις, το οίκης Ισλαμικό κράτος δηλαδή του Ιράκ και της Συρίας. Πρέπει να δούμε όμως ότι αυτές οι διαδικασίες δεν βοηθούν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των πραγμάτων. Ας ε, έχουμε μια πιο ε, μακροπρόθεσμη απάντηση που να βασίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της χάρτας των οικουμενικών δικαιωμάτων και να μπορέσουμε έτσι να ελέγξουμε την κατάσταση κλείνοντας και τις διάβλους για όπλα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κόσο Περμουή. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βαλέρο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα και στους οικείους τους τα θύματα της τρομοκρατικής απόπειρας ε, στο Παρίσι αλλά και παντού στον κόσμο. Πρέπει να καταπολεμηθεί φυσικά η τρομοκρατία. Σημαντικό είναι η πρόληψη, σημαντικό μέσο και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό. Κάνουμε λόγο για ένα ψήφισμα. Καλό και κακό αυτό. Ο πρόεδρος Ολάντα αποφάσισε να δρομολογήσει, να χρησιμοποιηθεί ρήτρα αμοιβαία συνδρομή εμείς. Είναι όμως πολεμικές δράσεις αυτές και κήρυξε τον πόλεμο στην τρομοκρατία όπως ο George W. Bush ε, μετά την 11η Σεπτεμβρίου από πλευράς Προεδρίας των ειπα και ακολούθησαν πόλεμοι. Γνωρίζουμε όμως ότι το αντίθετο επετεύχθη με αυτούς τους πολέμους και όχι η ειρήνη. Στο Παρίσι έχουμε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπεσαν θύματα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Δεν ήταν όμως επίθεση ενός ξένου κράτους. Το Νταέσο και στο Ισλαμικό Ισλαμικό κράτος Ιράκ και Συρίας ε, δεν είναι κράτος και αν θέλουμε να υπάρξει μια ρύθμιση ώστε να απαντούμε σε τέτοια εγκλήματα θα πρέπει να απαντούμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας με τα μέτρα ασφαλείας, δυνάμεις ασφαλείας, αστυνομία κτλ. Να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο άρθρο που να κάνει λόγο για την τρομοκρατία. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε λόγο για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Αλλά δεν θέλουμε να υπάρξει, να, να δοθούν διαστάσεις στην τρομοκρατία στην Ευρώπη δημιουργώντας μια στρατοκρατική κατάσταση, στρατοκρατοποιημένη κατάσταση και σε σχέση με το ψήφισμα αποφασίσαμε να καταθέσουμε ένα δικό μας κείμενο το οποίο αντανακλά καλύτερα τις αρχές μας και αξίες μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Στη συνέχεια ο συνάδελφος Χόκεν. Ευχαριστώ πολύ στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντα μα έλεγαν ότι δεν θα έχουμε στρατό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αλλά μετά τι επιθέσει των Παρισίων είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία που θα μπορούσε να έχει κανεί για το που κατευθυνόμαστε. Ακόμα και ο Τόνι Μπλερ τώρα ανοιχτά ζητά να τεθεί τέρμα στην εθνική κυριαρχία, δίνοντα τον έλεγχο του στρατευμάτων που έστειλε στον πόλεμο ε, στι Βρυξέλλε. Προσωπικά, όταν λέει ο Τόνι Μπλερ κάτι, ιδιαίτερα για το στρατό, η καλύτερη συμβουλή είναι να κάνει κανεί το αντίθετο Αντίθετα τον κύριο Μπλερ, εγώ, ε, θα, ε, εγώ είχα υποσχεθεί ε, πίστη στη Βασίλισσα όταν ήμουν στρατιώτη. Δεν μπορεί να βρείτε κανέναν που θα κάνει το ίδιο, να ορκιστεί πίστη στον κύριο Γιούνκερ. Έχουμε ήδη τι βάσει με τη ρήτρα αμοιβαία άμυνα. Αυτό θα συμβεί αν έχουμε και άλλη σύγκρουση όπου η Ευρώπη θα είναι διχασμένη. Τι θα γίνει αν η Αργεντινή με την υποστήριξη Τζέρεμι Κόρμπιν θέλει να, επισκεφ... επιτεθεί στα Φάουτλαντ ξανά θα σταματήσει τι πωλήσει αμυντικές και θα βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να υπασπιστεί τα νησιά. Ο πιο σημαντικό ρόλος οποιασδήποτε κυβερνήσεω είναι να προστατεύει τη χώρα τη. Γι' αυτό με την υποστήριξη τη συνθήκη τη Λαβώνας οι Ευρωβουλευτέ, του Ηνωμένου Βασιλείου έκαναν ζημιά. Διακόπτεται ο μιλητή. Ευχαριστούμε κύριε Χούκεμ. Για ένα λεπτό συνάρθος Όμπερμαερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω Αυστριακό είμαι υπερήφανο για την ουδετερότητα τη ε, χώρα μου και δεν δείχνω καμία κατανόηση όταν βήματα αναλαμβάνονται από τους αρχηγούς κυβερνήσεων αυτή η ε, ανεξαρτησία μας η στρατιωτική να υπονομευθεί και σε σχέση με την ε, ιδιότητά μας αυτή και ήδη με την δυνατότητα των τριών στρατηγικών ε, εταιρικών δεσμών που είναι σημαντική. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ότι για την Αυστρία είναι αυτονόητο το ότι συμμερίζεται αυτές τις αρχές Αυτά για την ανάλυση της κατάστασης ε, η ουδετερότητα όμως ε, και η διασφάλιση ε, ιδιομορφιών και ιδιωτήτων εθνικών είναι κάτι αυτονόητο ως θεμέλιο της Ευρώπης δεδομένης αυτής της κατάστασης. Και έτσι λοιπόν η ρήτρα συνδρομής δεν μπορεί να οδηγήσει με κανένα τρόπο στο να υπάρξει από, το παραπόρτι μια στρατιωτική συμμαχία η οποία θα υπονομεύεται κιόλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό παρακαλώ. κομμουνιστικό κόμμα της ελλάδας καταδικάζει το κοινό ψήφισμα που προβλέπει τη δημιουργία μόνιμου πολιτικοστρατιωτικού αρχηγείου επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 42 της ευρωσυνθήκης. τόσο η συγκρότηση αυτού του νέου στρατηγείου της ευρωπαϊκής ένωσης όσο και η ίδια ενεργοποίηση της λεγόμενης ρήτρας αμοιβαίας άμυνας σηματοδοτούν κλιμάκωση της υπεριαλιστικής επέμβασης στη συρία και στην ευρύτερη περιοχή με θύματα τους λαούς. αποτελούν ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της ευρωπαϊκής ένωσης στην κατεύθυνση συγκρότησης ευρωστρατού σε σύνδεση με το νατο ματοκυλάτε τους λαούς για το αν θα περάσει από τη συρία ο αγωγός του κατάρ σχέδιο των ηνωμένων πολιτειών και της ευρωπαϊκής ένωσης ή ο ρώσικος από το ιράν τα ίδια δεν κάνατε και στη λιβύη στο ιράκ και στο αφγανιστάν. τα προσχήματα και τα κηρύγματα αλληλεγγύης ηνωμένων πολιτειών ευρωπαϊκής ένωσης και νάτο και των κυβερνήσεών τους δεν πείθουν. τα υπερελιστικά σχέδιά τους έχουν και την ενεργή στήριξη της κυβέρνησης σύριζα ανέλ. ο ελληνικός λαός να εναντιωθεί στους υπερελιστικούς πολέμου απαιτώντας καμία εμπλοκή της ελλάδας σε αυτούς. ο πλούτος ανήκει στους λαούς αυτοί μπορούν και πρέπει να τον καρπώνονται. Ευχαριστούμε συνάδελφε Παπαδάκη. Ε, ακολουθεί ο συνάδελφος Μπροκ παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι αναπόφευκτη πράξη αλληλεγγύης να ακολουθήσουμε το αίτημα της Γαλλίας ώστε να, χρησιμοποιηθεί το άρθρο το οποίο επελέγει ως νομική βάση από αυτήν. Νομίζω ότι είναι και το ορθό άρθρο. Δεν θα ήταν ορθό να πάρουμε το άρθρο 5 της ρήτας συνδρομής του ΝΑΤΟ με μια αντιπαράθεση της δύση ε, και την ε, ε, Ισλαμική τρομοκρατία για το 122 για την τρομοκρατία στην εσωτερική, ε, στο εσωτερικό της Ένωσης αντί του εξωτερικού πρέπει να διαπιστώσουμε ότι είναι θέμα που αφορά τη συνεργασία όμως μεταξύ των κρατών μελών και όχι η ευρωπαϊκή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά το τι πρέπει να κάνουμε είναι το θέμα αν εδώ μπορούμε να δράσουμε με αυτόν τον τρόπο και να υπάρξει η σωστή συνεργασία και σε σχέση με παράδειγμα με τα, ε, την δύο ε, απάντησης από τα μέσα που διαθέτουμε κοινέ στρατηγικέ ε, πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε τι υπηρεσίε εκείνε για την διασφάλιση τη ασφάλειά μα και να μπορέσουμε στο κέντρο να δράσουμε άμεσα και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους μας σε σχέση με τον πόλεμο ο οποίος στην Μέση Ανατολή αν θα είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο για μας και η Εγγύς Ανατολή που πλήττεται από την τρομοκρατία με μια τελείως καινούρια διάσταση και έχουμε εδώ ε, θέμα επικράτειας, γεωγραφικής επικράτειας και βλέπουμε ότι υπάρχει μια νέα μορφή τρομοκρατίας με το Ισλαμικό κράτος και με τις κλασικές απαντήσεις του ΝΑΤΟ ΝΑΤΟ, δράσεις του ΝΑΤΟ, δεν έχουμε δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί εναντί αυτού του φαινομένου. Και πρέπει να δούμε σε σχέση με το επιτελείο και τη μόνιμη συνεργασία πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε πιο αποτελεσματικά και να μπορέσουμε να συνδράμουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόκ. Για δύο λεπτά η κυρία Γκόμες παρακαλώ στη συνέχεια η αμοιβαία συνδρομή που ζητείται από τη Γαλλία μετά από τα τελευταία πλήγματα τα τρομοκρατικά στο Παρίσι είναι πρόκληση να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις στην κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ας επισκεφθεί κανείς ε, τις πρώτες γραμμές στο Κουρδιστάν του Ιράκ για παράδειγμα τη σύγκρουσης ε, κατά του Ικής ε, και θα δει κανείς τι γίνεται με την Ευρώπη που δεν συνδράμουν τους πολεμιστές πεσμεργά των Κούρδων. Και αυτό παγκόσμια πρέπει να ισχύει. Απαιτούνται προσανατολισμοί ώστε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν συγκεκριμένες δράσεις για την αμοιβαία άμυνα. Χειροπιαστές δράσεις που θα συνεχίσουν ενώνουν ε, τα κονδύλια θα προασπίζονται τα στρατηγικά συμφέροντα επιβάλλοντας ε, τον κράτος δικαίου, rule of law. Αν δεν ξεπεράσουν ε, τις ανεδαφικές αρχές για την επικράτεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών τους οι ηγέτες μας και αν δεν περάσουν σε μια πραγματική πολιτική ασφάλειας και άμυνας που είναι ένα κλειδί για όλους για να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας Δημοκρατίας και παγκόσμια δεν θα είμαστε διαφορετικά αξιόπιστοι. Σας ευχαριστούμε και στη συνέχεια Φωτέγκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και μάλιστα προς μεγάλη έκπληξη πολλών βλέπουμε ότι μετά τις, ε, τα, ε, ε, τα τρομοκρατικά πλήγματα στο Παρίσι το άρθρο 42, εδάφιο 7 της συνθήκης ζητείται να χρησιμοποιηθεί και βλέπουμε ότι έχουμε εδώ ομόφωνα από πλευρά του Συμβουλίου ανταπόκριση για να συνδράμει την Γαλλία ομόθυμα και επιβεβαιώθηκε η θέση αυτή και φυσικά χρειαζόμαστε δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν μια ομόφωνη απάντηση του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και στη συνέχεια η κυρία Βάουτμαν θα λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπη, είναι η πρώτη φορά που ένα κράτος μέλος ε, το άρθρο 42 εδάφιο 7 επικαλείται για να λειτουργήσει και είναι αξιοπρόσεκτο ότι 27 κράτη ομόφωνα τοποθετήθηκαν θετικά υπέρ. Θα ήθελα να πω, δεν θα ήταν καλύτερο η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια να, να είχε επικαλεστεί αυτό το άρθρο για να υπάρξει μια αυθεντική από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης απάντηση, ομόθυμα. Δεν θα ήθελε να διευρύνει το Συμβούλιο αυτή τη διαδικασία ώστε να μπορεί το Συμβούλιο από κοινού με την Επιτροπή να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία. Δεν θα ήταν καλύτερο αυτό. Κυρία Μογκερίνη, είναι μια καταλητική ιστορικά στιγμή αυτή, καταλητική σημασία. Μετά από αυτά τα γεγονότα χρειαζόμαστε, πιστεύω, ένα ευρωπαϊκό στρατό, ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις που πρέπει να ε, ε, ε, οικοδομηθούν Λοιπόν, αν δεν το κάνουμε τώρα θα χάσουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στην συνέχεια η κυρία Σοφία Σακοράφα παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά έχουμε ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή. Υπόθηκε ότι δέχονται επίθεση οι αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση και η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Και επιβάλλεται αλληλεγγύη. Όλων. Προ όλου. Αμέριστη και απλόχερη. Γιατί οι ανθρώπινε αξίε δεν έχουν εθνική ταυτότητα. Όμως ποιο είναι ο εχθρός κύριοι συνάδελφοι. Οι κόλλες είναι οι άλλοι έλεγε ο Ζαν Πολ Σάρτ. Και αυτό είναι ο κίνδυνο. Ο τρόπο που υπερασπιζόμαστε τι ανθρώπινε αξίε να τι απαξιώνει και να γίνεται τροφοδότης αυτή τη κόλαση. Ποιο και γιατί βομβάρδισε και διέλυσε τι χώρε αυτέ και πνίγονται σήμερα χιλιάδε πρόσφυγε στη Μεσόγειο. Ποιο εξόπλισε του τζιχαντιστές υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι η υποχρέωση για παροχή στρατιωτικής βοήθειας και συνδρομής θα περιορίσει ή θα σταματήσει την κατάσταση αυτή. αλλαγή πολιτικής χρειάζεται κύριε συνάδελφε και κυρία μογκερίνη αλλαγή που θα αποκλείει πλήρως πολιτικές παρεμβάσεων και αποκλεισμών και θα κατευθύνεται αποκλειστικά στη χρησιμοποίηση μη στρατιωτικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό της φτώχειας την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την συμμετρική συνεργασία. ευχαριστώ ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ στα ελληνικά ο Πρόεδρος. Και στη συνέχεια η κυρία Ρίβαση παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Εγώ μετά από τη συγκίνηση των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων και τα συνηθισμένα ωραία λόγια, η ανικανότητα να καταπολεμήσουμε ξυλογικά την τρομοκρατία μας προλαβαίνει. Αυτή η ρήτρα αμοιβαίας ε, ε, συνδρομής 42-7 του Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται εξαιρετικώς και θέτει σε αμφισβήτηση μια πραγματική πολιτική κοινή άμυνας και κοινή ασφάλεια που πολλοί από εμά θα επιθυμούσαμε. Επιπλέον είναι εκτό θέματο γιατί οι τρομοκράτε που χτύπησαν τη Γαλλία προέρχονταν από την ίδια μα τη χώρα και αυτό θα έπρεπε να μα ανησυχεί. Οι λύσει εντό τη Ευρώπη για να καταπολεμήσουμε την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και τη συμβίωση. Εμείς εδώ δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, δεν συνδεόμαστε με τις αποφάσεις, κυρίως για αυτό το ε, άρθρο, ούτε καν η κυρία είπατε εκπρόσωπος. Αυτή η ρήτρα ε, στην ουσία σημαίνει την επιστοδρόμηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Διμερεί συνεννοήσεις μέσα στο πλαίσιο της, του κοινοτικού οικοδομήματος. Εγώ ως Γαλλίδα ε, που έχει αγωνιστεί για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας δεν καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιείται αυτό το άρθρο που είναι αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί στη συνέχεια η κυρία Αλιό Μαρή παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα στο όνομα του γαλλικού λαού να ευχαριστήσω καταρχάς όλες τις χώρες που προσέφεραν τη στήριξή τους σε αυτή τη ρήτρα θα ήθελα να του ευχαριστήσω βεβαίως για τα όσα ορισμένοι έκαναν πολύ συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα για το μήνυμα αλληλεγγύης που εστάλει σε αυτή την περίσταση. Ταυτόχρονα, κυρία Υπατή εκπρόσωπε, είναι αλήθεια ότι διάφορα ερωτηματικά για την εφαρμογή αυτής της ρήτρας θέτουν και το θέμα του κατά πόσο είμαστε, το, το τι μπορούμε να κάνουμε για να αμυνθούμε. Γιατί όλε οι χώρες, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να χτυπηθούν από την τρομοκρατία και ορισμένε ήδη έχουν χτυπηθεί και άλλε θα χτυπηθούν στο μέλλον δυστυχώ. Και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Ω πρώην Υπουργό Αμήνη, έχω δουλέψει εντό του ΝΑΤΟ και εκτό αυτού. Δεν είναι το ΝΑΤΟ η δομή που αντιστοιχεί σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται να υπερασπιστούμε τους συμπολίτε μας. Είναι η το πρώτο καθήκον ενός έθνους και ένα έθνος μόνο του αυτή τη στιγμή σήμερα δεν μπορεί να το καταφέρει. Όποιες και αν είναι οι δράσεις, όλες είναι διεθνείς. Δεν σημαίνει ότι καταλήγουμε την κυριαρχία μας, είναι θέμα πρακτικής οργάνωσης. Οπότε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε, όντως χρειάζεται να προχωρήσει η Ευρώπη της άμυνας. Πολύ συγκεκριμένα εσείς μας μιλήσατε, μας είπατε ποια είναι η σας για το θέμα αυτό. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή καταρχήν ενό γενικού στρατηγίου μονίμου. Χρειάζεται να προβλέψουμε και να μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα. Γιατί αυτό τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε εφόσον δεν υπάρχει ένα γενικό επιτελείο μόνιμο. Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ενότηση μέσα στη διαφορά ή διαφορετικότητα μέσα στην ενότητα. Δηλαδή πρέπει να αναπτυχθεί η μόνιμη δομημένη συνεργασία. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό είναι κάτι ρεαλιστικό και συγκεκριμένο. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, αναμένω τις απαντήσεις σας και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κυρία. Και στη συνέχεια Παρνιό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 13 Νοεμβρίου του 2015, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Φρανσουά Ολάντ, επικαλέστηκε το άρθρο 42-7 της Συνθήκης Σαββόνας στην ομιλία που έκανε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 Νοεμβρίου του 2015 έναντι της βαρβαρότητας και των φρικτών αυτών εγκλημάτων και της ε, επιθυμίας για θάνατο στην επικράτειά μας, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη ήταν η μόνη και μοναδική απάντηση. Σήμερα αυτή η αλληλεγγύη συμβολίζεται από αυτό το άρθρο, το 42-7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία πράγματι χρειάζεται μία αμοιβαία συνδρομή της Ευρώπης, διότι πολύ συχνά είναι μόνη της όταν καταπολεμά αυτούς που μας επιτίθεται. Πολλά κρατή-μέλη πολύ γρήγορα ανταποκρίθηκαν θετικά όσον αφορά την επίκληση των λόγω άρθρου. Χαιρετίζω αυτές τις αποφάσεις, τις αποφάσεις τους. Θα πρέπει λοιπόν να κοινοποιήσετε μια νέα παγκόσμια ε, γενική στρατηγική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Ιούνιο του 2016, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτή η επίκληση από πλευρά Γαλλία τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή να μπορέσει να λάβει μια επιχειρησιακή διάσταση. Πραγματικά είναι για πρώτη φορά που ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί αυτή τη ρήτρα. Λοιπόν, Ας ε, κάνουμε λοιπόν αυτή την κίνηση, ας ξεκινήσουμε ξανά το εργοτάξιο της Ευρωπαϊκής Άμυνας, κάτι που πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν. Δεν μπορούμε πλέον να κρυβόμαστε. Η Ευρώπη έχει προβλήματα ασφάλειας που είναι κοινά για όλα τα κράτη-μέλη ε, και αυτό στην άμεση γειτονιά της Ευρώπης συμβαίνει. Το Σαχέλ, εκεί Ανατολή, Μέση Ανατολή, είναι απλό το συμπέρασμα. Η ασφάλεια όμως είναι κοινή ασφάλεια, είναι περιφερειακή, δεν μπορεί να είναι κατακαιρματισμένη και διασκορπισμένη. Έναντι της καταστάσεως, μόνο μια πραγματική Ευρώπη της άμυνας θα ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία και η Γαλλία δεν θα μπορεί να ασχολείται μόνη της όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης. Ας μη φοβόμαστε λοιπόν να πούμε σε εκείνους που πάντα θέλουν λιγότερη Ευρώπη ότι σφάλουν. Και αντιθέτως, μοναδικά μέσω περισσότερης Ευρώπης θα καταφέρουμε να φτάσουμε να νικήσουμε και να πολεμήσουμε αυτή την τρομοκρατία σε αυτό τον πόλεμο που μας απασχολεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ιδού το εργοτάξιο, το πολιτικό, το πολύ σημαντικό που θα ξαναδώσει στην Ευρώπη ε, το, ε, το το, όλο, το ύψος, το κύρος που έχει χάσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου για την προσοχή σας και συνάδελφοι την προσοχή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική συζήτηση που θα πρέπει σήμερα ε, να τη συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο. Μαζί με σας να το κουβεντιάσουμε, μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τελικά να δώσουμε τις απαντήσεις που προσδοκούν όχι μόνο οι Γαλλίδες και οι Γάλλοι, αλλά τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί Λούκε παρακαλώ στη συνέχεια. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι απόλυτα σαφές ότι η Γαλλία <clears throat> την αλληλεγγύη, την υποστήριξη, την ενεργό βοήθεια όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αξίζει μια και απειλείται από την τρομοκρατία με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να βοηθήσουμε Ωστόσο οι πλειοψηφικές ομάδες σε αυτό το σώμα, οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες το χρησιμοποιούν αυτό ως ε, επιχείρημα για να δημιουργηθεί μια μονάδα άμυνας, μια κλίμακα πριν από την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού δεν είναι ορθό. Δεν χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκό Στρατό επειδή έπεσε θύμα τρομοκρατικών πράξεων η Γαλλία. Κυρίες και κύριοι συμβαίνει το εξής. Ένα σύστημα που να λειτουργεί το έχουμε με το ΝΑΤΟ για την άμυνα και ασφάλεια. Και με το ΝΑΤΟ πρέπει να αντιδρούμε αντιμετωπίζοντας κάθε απειλή στρατιωτική. Και μάλιστα σε σχέση με την Γαλλία, με την αλληλεγγύη, με την, τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχει η Γαλλία, πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος και τη συνδρομή τη δική μας. Όχι τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριο Ουρμπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, οι ε, τρομοκρατικέ πράξει στο Παρίσι ήθελαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα και ένα καθεστώ τρομοκρατία ε, στου πληθυσμού μα, ε, ανεγείροντα τύχη υποψίας και δημιουργώντα ένα καθεστώς έκθεση στη βαρβαρότητα. Και έτσι θα είχαμε απόλυτη νίκη τη τρομοκρατία, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι το ότι σε σχέση με το, ε, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν κατευθύνσει στρατοκρατικές όταν ο Μπούς για παράδειγμα στο παρελθόν ε, ανακήρυξε την διεθνή ε, εκστρατεία κατά το, του του τρομοκρατικού Ισλάμ, του Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Γι' αυτό απορρίπτουμε την ε, δράση ε, με βάση το άρθρο 42 εδάφιο 7 που θα μετατρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στρατιωτική συμμαχία. Ας καταπολεμήσουμε το φανατισμό και τη βαρβαρότητα και το φασισμό με περισσότερη δημοκρατικότητα και δημοκρατία χωρίς να εμπλακούμε στο εμπόριο μεταξύ δικαιωμάτων και ασφάλειας. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ευρωβουλευτά. Στη συνέχεια ο κύριος Μιλιάν Μον παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης κυρία Μογκερίνη για τα σχόλιά σας και τις επεξηγήσεις σας σε σχέση με το άρθρο 42 εδάφιο 7 και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Είναι αυτονόητο ότι η τρομοκρατική επίθεση που οδήγησε στο να λειτουργήσει ή να, γίνει επίκληση αυτού του άρθρου μας ε, θέτει όλους ε, ενώπιον της ε, τρομοκρατίας των συγχαντιστών. Και όταν συνήθανα άμεσα μετά από κάποιες μέρες μετά από τα τρομοκρατικά πλήγμα η οι Υπουργοί Άμυνα, αυτό έγινε. Έχουμε και υποχρεώσει ε, έναντι των εταίρων μα και έναντι των εταίρων του κόσμου, του αραβικού κόσμου. Έχουμε την μάχη κατά του, του Ντάεσ ε, και τη σύραξη στην ε, Συρία, τον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο όμω δεν επαρκεί η στρατιωτική απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζω ότι θα μπορέσει να προχωρήσει και να προοδεύσει παρόλη την αντίθεση που υπάρχει μεταξύ ε, ε, κάποιων κρατών. Αναφέρομαι στην κατάσταση στο Ιράκ, στο κέρα της Αφρικής. Οι δικές μας δράσεις πρέπει να στρέφονται υπέρ του, της προστασίας των γειτόνων μας και των συμμάχων μας. Βλέπουμε ότι υπονομεύεται η διεθνής ασφάλεια και στο τέλος τέλος η δική μας ευρωπαϊκή ασφάλεια και ολοκληρώνω με ένα τελευταίο σχόλιο. Οι διάφορες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή επικράτεια και σε σχέση με τις σειράξεις στη γειτονία μας είναι ένας λόγος για να προχωρήσουμε στην εμβάθυνση όπως αναφέρθηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη δρομολόγηση των διαφορετικών μηχανισμών που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο Πίκουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Μετά τις ε, τρομοκρατικέ πράξει στο Παρίσι πέρσι, ο Γάλλο Υπουργό Άμυνα, για πρώτη φορά στην ιστορία αναφέρθηκε στην επίκληση του άρθρου 42 εδαφίου 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λόγω τη ένοπλη αυτή επίθεση κατά τη Γαλλία. και ζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν. Πολλοί ερμηνεύουν αυτό το τμήμα τη συνθήκη Λισαβόνα σαν ένα είδο παραρτήματος στο άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ε, σύμφωνα με το οποίο όταν υπάρχει επίθεση κατά ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν. Δεν μπορούν να, να αμελήσουν αυτό το αίτημα της Γαλλίας οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να μπορέσει να βοηθηθεί η Γαλλία πολύτροπα και πολυσχηδώς και όχι υποχρεωτικά μέσα σε ένα στρατιωτικό αποκλειστικά πλαίσιο. Είναι θέματα και της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και το καλύτερο θα ήταν εδώ σε αυτή την περίπτωση η ε, εξωτερική πολιτική να μην είναι ο πιο ευάλωτος κρίκος ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το 2014 γίναμε μάρτυρες όλοι του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα σύστημα ενιαίο σύστημα άμυνας θα μπορούσε να εξοικονομήσει πάρα πολλά χρήματα. Δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως ε, αληθεύει ότι δημιουργούνται πολλές φορές ερωτήματα περισσότερα από τις απαντήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ομοιογενής τρόπος αντίδρασης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια ε, θα λάβει τον λόγο Μπαρεκόφ. Ευχαριστώ. Υπάρχει ο τρόμος διότι κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να περάσει τα σύνορα. Όχι διότι δεν έχουμε ευρωπαϊκό στρατό, κάποιος θα πρέπει να υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα διότι η ειρήνη κινδυνεύει. Η μέθοδοι των ζόμπι του Ντάες είναι απειλή κατά των ευρωπαϊκών χωρών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν ένα πόλεμο ο οποίος απαιτεί μεγάλα μέσα. Η χώρα μου είναι εξωτερικό σύνορο, όμως η χώρα μου είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Όμως πρέπει να έχουμε τα μέσα που θα ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων. Η χώρα μου είναι θέατρο επιχειρήσεων και μάχης μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αντί να δημιουργηθεί ένα επιτελείο, ένα αρχηγείο, θα πρέπει η Ευρώπη να μας δώσει τα μέσα για να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια η κυρία Κανιέτε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, Αντιπρόεδρε, η σημερινή μας συζήτηση είναι μια σκληρή υπενθύμηση ότι έξι χρόνια μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε ακόμα ρυθμιστικές, ε, ε, μάλλον ε, ρυθμίσεις εφαρμοστικές όπου η συνθήκη έχει μείνει συμβολική και πολιτική παρά πρακτική. Αντίθετα με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει κάποιο συνδυασμό και κάποια δομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή αυτού του άρθρου της της Η απάντηση στις επιθέσεις στο Παρίσι και οι εξελίξεις των περασμένων ετών απέδειξαν ότι χρειάζεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση Αμήνης που θα περιλαμβάνει τις χώρες που θέλουν να ε, συνεργαστούν στενότερα σε αμυντικά θέματα και θέλουν να προχωρήσουν με αστυνομική βάση μόνιμη και οργανωμένη συνεργασία. Χρειάζεται επίσης μόνιμο γενικό επιτελείο με σχεδιασμό για συλλογική άμυνα και στη στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ασθενοτερη συνεργασία Ένωση ΝΑΤΟ είναι βασική για την υπεράσπιση των κρατών μα, των κοινωνιών μα και των δομών μα στο μέλλον. Δεν χρειάζεται να ξαναεφεύρουμε το τροχό, αλλά να, ε, να οργανωθούμε για κάθε είδου επίθεση. Είτε παραδοσιακέ στρατιωτικού τύπου, είτε ε, πιο ε, εξυγχρονισμένε. Εδώ η Ένωση πρέπει να παίξει βασικό ρόλο. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε. Όπως ξέρετε είναι η πρώτη φορά όπου επικαλείται κάποιο κράτος σε την ρήτρα αμοιβαίας αρρωγής. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα και να αναπτύξουμε συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές που θα μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στο μέλλον. Για να ενισχύσουμε τη συνεργασία στα θέματα πληροφορίας και συνεργασίας. Είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι συλλογικά δαπανούμε πολύ περισσότερα χρήματα ο καθένας μας για την ενώ συλλογικά όχι, γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι μας διαφεύγουν οι τρομοκράτες επειδή δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Πώς ε, θα δεχτούμε ότι αποτυχάνουμε τον έλεγχο ε, πωλήσεων στη μαύρη αγορά. Η ευρωπαϊκή συνεργασία σημαίνει, είναι η απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε την κυριαρχία ή ότι θα καταπατήσουμε ή θα βάλουμε στην άκρη τον Άντο. Σημαίνει το 42-7 το να είμαστε έξυπνοι, να στηρίζουμε τις συνεργασίες, να ε, κάνουμε κοινά έρευνες, προμήθειες και να αυξάνουμε την ολοκλήρωση του εισαγοράς. Εγώ καλώ το Συμβούλιο να καταστήσει αυτό το ζήτημα προτεραιότητα. Κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσανέσκη, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, κυρία Μογγελή. Μετά από τις ε, φρικαλές ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, η Γαλλία αποφάσισε να επικαλεστεί αυτή την ε, ρήτρα αμοιβαία άμυνα του άρθρου 42 παραγράφου 7 τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά και με αυτό τέθηκε σε δοκιμασία η προετοιμασία, η ετοιμότητα των κρατών μελών να ανταποκριθούν με τα όσα προβλέπει η συνθήκη άμεσα. Το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι διμερώς να υπάρξει η δραστηριοποίηση και είδαμε ότι υπήρξε υψηλή δέσμευση ολόκληρη σειρά κρατών μελών να βοηθήσουν τη Γαλλία διμερώς και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι άλλες στρατιωτικές δράσεις στις οποίες συμμετέχει η Γαλλία και που σίγουρα θα πρέπει να προσαρμόσει βελτιώσει την παρουσία της αντίστοιχα. Πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί συνεργασίας, διαρκούς συνεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με μια ολόκληρη σειρά προσπαθειών που ε, ε, εσείς ε, εξετάσατε και αναφέρατε κυρία Μογκερίνη και που εντάσσονται στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας και μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και στο άρθρο του 5 του ΝΑΤΟ και το 222 και το άρθρο 42 ε, παράγραφο 7 πρέπει να δούμε μεταξύ όλων αυτών των δυνατοτήτων πώς μπορούμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι στην προάσπιση της άμυνάς μας. Εδώ εντάσσεται και το λευκό βιβλίο για την άμυνα που αποτελεί μία από τις προτεραιότητες ε, για εμάς τους επόμενους έξι μήνες και την ε, επόμενη Προεδρία επίσης. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια Ζάλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ψήφισμά μας σωστά ζητά ε, ασφάλεια και εγγυήσει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισότιμα. Και σωστά το ψήφισμά μας ζητά ε, να υπάρχει θέση Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε και το άρθρο 42.7 της συνθήκης που επικαλείται η Γαλλία. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν πρόβλημα μόνο διμερός. Τα αιτήματα αυτά, οι εγγύησει για την ασφάλεια των πολιτών και η έδρα, η θέση, η έδρα του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ, όλα αυτά μπορούν να βρουν απάντηση να έχουμε ένα ευρωπαϊκό επιτελείο και κοινό ευρωπαϊκό στρατό, έναν μικρό επιχειρησιακό στρατό που θα είναι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο αυτό, χρειαζόμαστε και Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Πληροφοριών Χωρίς αυτούς τους δύο φορείς, το κοινό επιτελείο και ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες, ευρωπαϊκή μυστική υπηρεσία μάλλον, ε, δεν θα μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες που προανέφερα. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Κέλαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μογκερίνη, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την Ισλαμική τρομοκρατία θα πρέπει να είναι ένα κοινό νέο πρόγραμμα για όλους τους πολίτες και όλα τα κράτη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη και αμοιβαία συνδρομή για την αμοιβαία άμυνα τα τρομοκρατικά πλήγματα στη Γαλλία ήταν καταλήτης ε, ώστε να επικαλεστεί η Γαλλία την ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, αμοιβαία άμυνας μέσα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Πρόκειται για τις εντάσεις που υπάρχουν, το πεδίο εντάσεων όσον αφορά την ίδια την ασφάλειά μας. Αυτό όμως το δυναμικό το οποίο έχουμε είναι μάλλον περισσότερο θεωρητικό δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Τίθεται το ερώτημα αν με το άρθρο 222 θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από με το άρθρο 42 παράγραφο 7 ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και όλα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα λοιπόν αυτό να ενδυναμωθούμε, να ενισχυθούμε από κοινού με το ΝΑΤΟ να ενισχύσουμε και να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και αν ένα μέρος ενός κράτους υφίσταται επίθεση από τους τρομοκράτες να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Μία, ένα άλλο επιπλέον τελευταίο συμπέρασμα. Το δυναμικό το οποίο έχουμε για να το χρησιμοποιήσουμε χρειαζόμαστε ένα κεντρικό επιτελείο στρατηγικού χαρακτήρα και ε, στρατιωτικού χαρακτήρα. Πρέπει να υπάρξει αυτή η πρόνοια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια πρέντα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που αγρίως χτύπησαν την Γαλλία δεν χτύπησαν μόνο τους Γάλλους αλλά όλους τους Ευρώπους. Η μόνη και δυνατή δράση για να καταπολεμιστεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία θα πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή λύση. Η ρήτρα αμοιβαία ε, συνδρομής είναι μια πρώτη φάση και πρόκειται για μια βάση στην υποχρέωση αλληλεγγύης που είναι επίσης μια ισχυρή ε, ε, πολιτική δράση απέναντι σε αυτή την ε, τρομοκρατική απειλή. Πολλές χώρες απάντησαν θετικά στο αίτημα της Γαλλίας και θέλω να χαιρετήσω τη γρήγορη αντίδραση και τη δέσμευση ορισμένων κρατών μελών. Η πραγματική επένδυση των ευρωπαϊκών χωρών είναι φυσικά πολύ διαφοροποιημένη και θα πρέπει οι προϋποσχέσεις να ακολουθηθούν από συγκεκριμένες δράσεις. Αλλά ακόμα και αν οι μεμονωμένες συμβολές ε, δεν μπορεί να είναι να είναι περιορισμένες, αν τις προσθέσουμε δεν είναι καθόλου ομελητές. Η δραστηριοποίηση αυτής της ρήτας προσφέρει εξαιρετικό παράθυρο ευκαιρίας για να ενισχυθεί η πολιτική αμήνης και ασφάλειας. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ορίσουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική σε θέματα αμήνης, να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και τα μέσα μας δεν είναι επιλογή πλέον, είναι απόλυτη ανάγκη. Δεν μπορεί ο καθένας να ενεργεί μόνος του, ανάλογα με τις πεπιθήσεις και τις προτεραιότητές του. Οι προτεραιότητες είναι πλέον κοινέ. Η καταπολέμηση του ΤΑΕΣ, να τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία, να σταθεροποιηθεί η Λιβύη. Η Ένωση πρέπει να ενεργήσει ως ένας, ε, ένα μπλοκ για να σημάνει τη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Μαγκερίνη, οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν λύσεις γρήγορες και αποτελεσματικές, διότι ήδη εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να βοηθά ανάλογα με τις δυνατότητες. Εμείς μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία, τη ΣΥΠΑ, τα αραβικά κράτη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στα πλαίσια τα θεμητά θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ε, μελλοντικά την ειρήνη στο Ιράκ και τη Συρία, ούτως ώστε οι μετανάστε ε, που βρίσκονται στην επικράτειά μα σήμερα μπορούν να επιστρέψουν. Κυρία Μογκερίνη, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ενεργοποίηση του άθρος 42-7 ω καταλήτη πριν, για να δημιουργήσουμε δυνατότητα, δυναμικό ασφάλεια και άμυνα Ευρωπαϊκή Ενώσεω, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών και ευρωπαϊκού στρατού. Σαν πρώτο βήμα γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κέντρο πολιτικό και στατιωτικό σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο που θα συντονίζει τα διάφορα σχέδια δράσεως σε περίπτωση κατεπίγουσας ανάγκης και άλλες επιχειρήσεις που θα πορεύουν την ενεργοποίηση του 42 42-7. Πρέπει να υπάρχει μόνιμη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη με τις δομές του ΝΑΤΟ. Για να επιλύσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα όπως η μετανάστευση, η καταπολέμηση τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ντροπή που οι ηγέτες της Βρυξέλλες παίρνουν αποφάσεις αλλά δεν ε, ανταποκρίνονται μέσω οικονομικής ε, ενίσχυσης να πετύχουν τους στόχους. Ευχαριστώ στη διαδικασία τώρα Catch the Eye. Πάμε. Ο κ. Μάσιτς έχει το λόγο. Κυρία Μάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω, πρέπει να πω, <clears throat> ότι με αυτή την τρομοκρατική απειλή πιστεύουμε και θεωρούμε όλοι ότι δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με ένα από πλευρά ενό κράτου μόνο. Χρειάζεται συντονισμένη δράση και στοχοθετημένη δράση. Και η αμοιβαία άμυνα, όχι μόνο σύμφωνα με το 42-7 ε, τη ε, ε, συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή πρόκειται για την προάσπιση των συμφερόντων μα. Δεν, δεν έχω τη βεβαιότητα ότι αυτό το άρθρο είναι ο καλύτερο τρόπο για να το κάνουμε αυτό ε, μόνο ε, ε, αν ήταν θύμα μιας στρατιωτικής δράσης η Γαλλία θα μπορούσαμε να το κάναμε. Αν το κάνουμε χωρίς να έχει υποστεί μια στρατιωτική επίθεση τότε θα ωφεληθούν οι Ισλαμιστές. Και αυτό σε σχέση με παρόλες τις προσπάθειες των τρομοκρατών να εμφανίζονται ως κράτος πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα τρομοκρατικά πλήγματα ως τρομοκρατικά πλήγματα απλά και ξεκάθαρα. Και γι' αυτό η επίκληση του άρθρου για την αμοιβαία συνδρομή δεν είναι το πιο επαρκές μέσο. Παρότι αυτό βέβαια δεν παρακολεί αν επιθυμούν τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν έστω και στρατιωτικά τη Γαλλία. un minuto per favore. Grazie Presidente, ottimo Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιρετικά τα Ιταλικά σας. Ε, το αίτημα της γαλλικής ε, κυβέρνησης να επικαλεστεί τη ρήτρα αμοιβαίας αρρωγής το 42-7 τουλάχιστον ε, επί της αρχής αποτελεί μια ευκαιρία αλλά ίσως και μια χαμένη ευκαιρία και από δικονομικής άποψης. Από αυτή την άποψη το άρθρο 222 που ορίζει την περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος πέσει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης ίσως θα ήταν καλύτερο να το επικαλεστεί. Το ίσως δεν μπορεί να θεωρηθεί όντω κράτος. Ε, ε, ε, ε, Πάντως δεν θεωρείται, δεν το έχουμε εμεί αναγνωρίσει. Έπειτα αυτή η επιλογή ε, διακυβερνητική μέθοδο έναντι της ε, της κοινοτικής και διάφορα κράτη χρειάστηκε λοιπόν έτσι να κληθούν να βοηθήσουν. Ωστόσο η Ευρώπη δεν συμμετείχε, δεν μπόρεσε να δώσει μια συντονισμένη απάντηση. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία για να αποδείξουμε την Ευρωπαϊκή Ενότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, η ρήτρα αμοιβαία άμυνα που ορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης και άρθρο 222 συνθήκης λειτουργίας ευρωπαϊκής ένωσης ορίζει ρητά ότι οι δράσεις υποστήριξης ενός κράτους μέλους που έχει δεχτεί τρομοκρατική επίθεση αφορούν αποκλειστικά και μόνο το έδαφος του μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών. τονίζουμε λοιπόν ότι η ρήτρα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας κανενός κράτους συνεπώς το αίτημα της γαλλίας για υποστήριξη στρατιωτικών αποστολών σε αφρική και μέση ανατολή είναι νομικά αβάσιμο. ας σημειωθεί εδώ ότι οι στρατιωτικές αυτές αποστολές στην καλύτερη περίπτωση είναι τυχοδιοκτικέ και ουδόλως συνδράμουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας όπως ξεκάθαρα φάνηκε στην συριακή κρίση το. 2011. άλλωστε όπως τονίζει έρευνα ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης που επιβεβαιώνουν διαρκώς πληροφορίες που διαρρέουν στον τύπο πέραν του νταές ένα μεγάλο μέρος της συριακής ένοπλης αντιπολίτευσης που υποστήριξε θερμά η γαλλική δημοκρατία αποτελείται από ομάδες ισλαμιστών πράγμα που δείχνει το ποιόν των συγκεκριμένων οργανώσεων και το ότι δήθεν το αγνοούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. τα κράτη μέλη οφείλουν να μείνουν μακριά από εξωτερικές επεμβάσεις και υπεριαλιστικούς πολέμους. ευχαριστώ. Ε, ε, Κύριος Επιτίδιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, αποτελεί μια υψηλού επίπεδου δέσμευση των κρατών μελών να στηρίξουν ένα άλλο κράτος το οποίο είτε δέχεται αμέσως επίθεση στο έδαφος του είτε απειλείται με μελλοντική στρατιωτική προσβολή. αυτή είναι μια πολύ ωραία απόφαση η οποία υπονοεί την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ενώσεως να επιδείξει αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη της. πόσο όμως πραγματικά πιστεύουμε σε αυτή την περίπτωση. εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά πω η τουρκία απειλεί την ελλάδα ένα μέλος της ευρωπαϊκής ενώσεως με πόλεμο κάζο μπέλι εάν ασκήσει νόμιμα δικαιώματά του. επίσης η τουρκία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ενό άλλου κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ενώσεως της κύπρου και την απειλεί ανάλογα. ποια είναι η στάση την οποία έχει επιδείξει η ευρωπαϊκή ένωση απέναντι σε αυτή την προσβολή; έχει απαιτήσει από την τουρκία να πάψει να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο; και αν σε αυτή την απλή περίπτωση δεν έχει επιδείξει αποφασιστικότητα η ευρωπαϊκή ένωση πώς περιμένουμε να επιδείξει αποφασιστικότητα όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και απαιτούν στρατιωτική επέμβαση. Ομπριγάδο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ στα ελληνικά. Και τώρα η κυρία Μογκερίνη θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ η Επίτροπο. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ σαφώς αντιμετωπίζουμε ένα είδος απειλής που παλιότερα, μόλις πριν από έξι χρόνια στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας δεν είχε προβλεφθεί γιατί ε, όταν πρόκειται για εσωτερική απειλή, ας θυμόμαστε πάντοτε ότι η εθνικότητα των τρομοκρατών ήταν ε, ευρωπαϊκή αλλά με σαφή εξωτερική σύνδεση γιατί υπήρχε σύνδεση, υπήρχε κατάρτιση, πόρη, στήριξη που το συνέδε με τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και με τον ΤΑΕΣ. Σαφώς λοιπόν η γραμμή ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική απειλή, ακόμα και μόλις πριν 6 χρόνια, ήταν πολύ καλύτερα καθορισμένη από ό,τι σήμερα. Η φύση της απειλής λοιπόν, και αυτό θα θέλω να υπογραμμίσω, είναι επίσης για προσαπάντηση ορισμένων από εσά που αναφέρθησαν στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Θυμηθείτε παρακαλώ ότι η επιθέσεις στο Παρίσι δυστυχώς διαπράχθησαν από ανθρώπους που είχαν ευρωπαϊκά διαβατήρια. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα υπεράσπισης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής από εξωτερικές απειλές, αλλά είναι και το πολύ πιο περίπλοκο ζήτημα του πώς θα ασφαλίσουμε τους πολίτες μας, πώς θα εγγυηθούμε την ασφάλεια των συμπολιτών μας από, από τις απειλές που ταυτόχρονα είναι εσωτερικές και εξωτερικές. Και πρέπει να συνδυάσουμε διαφόρων ειδών μέτρα. Πιστεύω και ελπίζω ότι η γενική η στρατηγική επί τη οποία εργαζόμαστε θα μας βοηθήσει να επανακαθορίσουμε μια κοινή κατεύθυνση και για το πώς θα εγγυηθούμε την ασφάλεια των συμπολιτών μα Για αυτού του καιρού, αυτούς τους δύσκολους καιρού, νέες απειλές ε, που είναι πολύ διαφορετικές. Τούτο λεχθέντω θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία που αναφέρατε. Πρώτον, χρήση του άρθρου 42.7 αντί του 222. Βεβαίως, καταρχήν, το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει την πολιτική απόφαση για το ποιο άρθρο θέλει να επικαλεστεί όταν ζητά την αρρωγή των άλλων κρατών μελών. Θα ήθελα να συγκρίνω τα δύο άρθρα. για το οποία συζητάμε εδώ. Το 42.7 αναφέρεται σε ένοπλη επίθεση ή ένοπλη ε, ε, σύραξη. Έχουμε διαφορετικές ε, διατυπώσεις στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές και το άρθρο 222 ε, αναφέρεται σε τρομοκρατική επίθεση ή τρομοκρατική καταστροφή. Και στις δύο περιπτώσεις τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν Όσον αφορά τη συμβολή του στην περίπτωση του 42-7, η βοήθεια προέρχεται από τα μονομένα κράτη-μέλη ενώ ορισμένοι από εσάς υπογράμμισαν ότι το 222 ζητά καλή μάλλον και την κινητοποίηση ευρωπαϊκών μέσων. Όσον αφορά την εφαρμογή, και εδώ νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις, το άρθρο 42 42F7 αφήνει τη διαδικασία εφαρμογής ανοιχτή και εδώ μπορώ να παρατηρήσω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που εσείς υποδεικνύετε θα ήταν χρήσιμες για το 2012. Αλλά σήμερα διαπιστώνουμε την εφαρμογή αυτού του άρθρου, όταν δηλαδή συγκεντρώσουμε τους πόρους μας, τις υπηρεσίες μας, τις συμβουλές μας. Αυτό είναι που κάναμε. ανάμεσα στην λήψη της απόφασης με την γαλλική κυβέρνηση να χρησιμοποιηθεί το 7-7 και τη στιγμή που έγινε το Συμβούλιο ε, με τους Υπουργούς Αμήνης. Σε 24 ώρες δηλαδή μπορέσαμε να συγκαλέσουμε το Συμβούλιο Αμήνης. Και πιστεύω ότι η δουλειά που έκανε η νομική μας υπηρεσία και η δομές μας και προσέφεραν αυτό το επίπεδο βοήθεια ήταν πολύ θετικό. Και ο συντονισμό των κρατών μελών, αλλά και πάλι για το εφαρμοστικό άρθρο 222, εκεί λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντονιστικό ρόλο να παίξει λόγω της δυνητικής ε, εμπλοκή ε, ευρωπαϊκών μέσων. Ακόμα και αν η διατύπωση του 42-7 δεν απαιτεί συγκεκριμένο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα εφαρμογής, εμείς αποφασίσαμε από κοινού με τη Γαλλία και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στη διάρκεια του Συμβουλίου εκείνου της 17ης Δεκεμβρίου να εμπλακούν άμεσα εμού συμπεριλαμβανόμενη στην όλη διαδικασία ε, και όλα τα ευρωπαϊκά ε, μέσα και όργανα. Και αυτό δείχνει την προθυμία μας να χρησιμοποιήσουμε αυτό το άρθρο ως έναν τρόπο να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, αυτή την, σε αυτό το τομέα. Ένα στοιχείο μπορεί να σας φαίνεται τεχνικής αλλά εγώ πιστεύω πως είναι σημαντικό. Το ανέφερε ο Έλμαρ Μπρόκ η τοποθεσία της δράσης. Ε, αφορά διαφορετικά μέρη, το 42.7 και το 222. Για το 42.7 η βοήθεια δίνεται εντός της επικράτειας του κράτου μέλους για να ενισχύσει τις δυνατότητες του, τις ικανότητες του στη διάρκεια κρίσης, ενώ στην περίπτωση, συγγνώμη, το 222 είναι αυτό, ενώ στο 42-7 σαφώς επρόκειται για βοήθεια σε εξωτερική ε, δράση, εξωτερική επικράτεια. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο που σαφώς ελήφθη υπόψη. Υπήρχαν και άλλα άρθρα που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός από αυτά τα δύο, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε και το άρθρο 44 που δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, ούτε και αυτό. Και αυτό θα σήμαινε δράσεις της ΚΕΠΑ και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Με τα πρόθυμα κρατημέλη, λέει το άρθρο, αν, το, το θυμάμαι καλά, που αναλαμβάνουν την ευθύνη, κοινού με το Συμβούλιο να ε, προβούν σε μια επιχείρηση ΚΕΠΑ ε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου πολιτική θέση είναι και φαντάζομαι πως το Συμβούλιο θα ε, στηρίξει αυτή μου τη θέση ότι δεν θα ήταν σωστό, δεν θα ήταν πρέπον η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια να προβεί σε ε, στρατιωτική επιχείρηση κατά του ΤΑΕΣ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή, όχι τεχνική χρήση των συνθήκων. Και πιστεύω και ότι και εδώ στο ημικύκλιο οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι για την ώρα τουλάχιστον μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια θα έπρεπε να προβεί σε μια επιχείρηση στρατιωτική κατά του Ντάις στο Ιράκ. Γιατί, γιατί έχουμε άλλες δυνατότητες συμμετοχή τη ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα. Την επόμενη λες, ναι. Στην ε, φάση τη εφαρμογή του 42.7, στην ουσία πρόκειται για αναβάθμιση των θεσμών της Ένωσης σε σχέση με τη διατύπωση του άρθρου και από την άλλη πλευρά το αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε τη διπλωματική και ανθρωπιστική εργασία, καθώ και την εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντό του Συμμαχίας κατά του ΝΤΑΕΣ, εφόσον έχουμε δεσμευτεί και παγκοσμίω κατά του ΝΤΑΕΣ. Τώρα, για το ΝΑΤΟ. Για τα κράτη-μέλη που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ, η αμοιβαία αρρωγή τη Ένωση είναι συμπληρωματικό στοιχείο στην συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και αυτό σαφώ αναφέρεται στο άρθρο 42.7 που λέει ότι οι δεσμεύσει και η συνεργασία σε αυτό το τομέα θα είναι σύμμορφα με τις δεσμεύσει ε, που απορρέουν από την ε, συνθήκη τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Καμία κανείς συμπληρωματικέ είναι οι δράσεις. Και να πω και γενικότερα ότι εμείς ενισχύσαμε αυτό, σε αυτόν τον χρόνο και κάτι που έχουμε αναλάβει υπηρεσία. Εγώ ως είπατε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύριος Στόλτεμπεργκ ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ένωση σε πολύ μεγάλο βαθμό και αναμένω ε, ότι θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερη συνεργασία μας καθώς αναπτύσσουμε τη στρατηγική μας και καθώς το ΝΑΤΟ προετοιμάζει την διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Οι δυο διαδικασίες προχωρούν παράλληλα και βεβαίως ε, ε, έχουμε τελείως διαφορετικά μονοπάτια, αλλά επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδιαίτερα για τους τομείς όπου η συνεργασία μας μπορεί να είναι παραπληρωματική και προς όφελος όλων, όπως για παράδειγμα στους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να προσθέσει αξία. Υπάρχουν τομείς συνεργασίας δηλαδή που προχωρούν. Να πω επίσης ότι η γαλλική απόφαση να επεκαλεστεί το 42-7 ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και θα έπρεπε να θεωρηθεί ως ένας αποτελεσματικός προμηθευτής ασφάλειας. Πρώτα απ' όλα από τα ίδια της τα κράτη. Δεύτερον ότι η αλληλεγγύη είναι κομμάτι της Ένωσης. Ότι όλα τα άρθρα της συνθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και να σας πω επ' αυτού ότι δεν χρειάζεται να γίνουν ιδεολογικές θεωρητικές συζητήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις σε αυτή τη φάση που η ασφάλεια της Υπήρου μας ε, είναι υπό επίθεση. Δεν χρειάζεται θεωρητική συζήτηση, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να δημιουργήσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις για να το κάνουμε αυτό, τονίζοντας την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης και στη διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας, όπου μπορεί να είναι ένα πολύτιμο και ζωτική σημασία σε εργαλείο προς την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων σε ορισμένε περιπτώσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσθεθέμενη αξία γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε 17 αποστολές και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο ήδη που είναι μέσο και εργαλείο ε, που, ε, όπου λειτουργούν όλα τα κρατημέλη μαζί, που ενεργούν μαζί, γιατί όλοι μαζί είμαστε καλύτεροι από ότι ο καθένας μόνος μας. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου τα ευρωπαϊκά μέσα ήταν καλύτερα από ότι τα ε, νατοϊκά ή τα μέσα, οι αποστολέ του ΟΗΕ. Και αυτό είναι κάτι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ορμόφωνα αναγνωρίζει στα πορίσματά του του Δεκεμβρίου και του, του 13 και του Ιουνίου 15 υποδεικνύουν μια κατεύθυνση που τονίζει τη διάσταση της, ε, της ΚΕΠΑ. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι Πρέπει να προετοιμάσουμε πολιτικά την, αυτή την υπόθεση ώστε να επιτύχουμε την εφαρμογή των διατάξεων των συνθήκων πλήρως και επιτυχώς υπέρ της ασφάλειας και προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μογκερίνη. Και έτσι ολοκληρώθηκε